Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρία σε με έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ζήθηκε να αναβληθεί το σημείο 8 για το εμπόριο της μπανάνας για αύριο μετά το σημείο 21. Επίσης ζητήθηκε να γίνει πιο νωρίς η ψηφοφορία για τα δικαιώματα του ανθρώπου και κοινωνικέ προδιαγραφέ και προδιαγραφέ περιβάλλοντο για τι διεθνεί επιστημονικέ. Ε, Εμπορικέ συμφωνίε συγγετή Κασμαρέκ προβλέπεται για αύριο, σημείο 14. Να το συζητήσουμε δηλαδή σήμερα στι 18 ε, και 15, μετά το σημείο 10. Επειδή ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή εμπορίου προβλέπεται για αύριο το πρωί. Για τα σημεία 16 για την διάσκεψη Αφρική Ένωση δεν θα ψηφίσουμε μέχρι να συνεδράσουν οι συντονιστές αύριο το πρωί. Ωστόσο η συζήτηση θα γίνει όπως προβλέπετε σήμερα. Αντιρρήσεις ή σχόλια. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η μυρίσια η μυρισια και με αυτές τις αλλαγές. ώρα των ερωτήσεων. Είχα κάνει μία ερώτηση προς την Κομισιόν 2 Ιουνίου του 2010 για ένα σχέδιο ανάπτυξης στην Αγκόλα Agri International. Κακώς αποδόθηκε στην κυρία Κέλλα και στον κύριο Μπέρμαν η ερώτηση. Τεχνικό λάθος. Εγώ είχα κάνει την ερώτηση. Παρακαλώ την Κομισιόν να απαντήσει. Είναι πρόκειται για την συνέχεια δραστηριότητας για τη μη κυβερνητική οργάνωση Αγκρεσίντε. Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ο Αρμόδης δεν έχει έρθει ακόμη. Από μια ανταλλαγή email συνάγω ότι το αίτημα της Αγκρεσουίντ το συζητάνε οι Ευρωπαίοι διαμεσολαβητές και το αξιολογούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να σας δώσουμε επιπλέον πληροφορίες. Ενώ δεν έχουν αποφασίσει οι μεσολαβητές. Που μπορεί να είναι η απόφαση του είτε υπέρ της Κομισιόν είτε υπέρ της Αγκρισίδ. Αν υπάρξει πρόβλημα κακοδιαχείριση εκ μέρου των υπηρεσιών τη Κομισιόν, αν αποδειχθεί αυτό. Δυστυχώ, δεν μπορώ να σα πω τίποτε παραπάνω. Προέδρο. ευχαριστώ. Έχει να μας κάνει καμία ανακοίνωση η Κομισιόν. Όχι. Οπότε ερχόμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Γεωργικές τεχνολογίες για αναπτυσσόμενες χώρες. Παρουσίαση του σχεδίου στο ΣΤΟΑ. Προσκαλέσαμε και Χαιρόμαστε γιατί έχουμε εδώ τον κύριο Πολ Ρεμπίκον, πρόεδρο τη Επιτροπή στο Κοινοβούλιο μα για την αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων. Στο είναι τα αγγλικά αρχικά Scientific and Technological Options Assessment. Όπως ξέρετε η ΣΤΟΑ είναι το πλαίσιο αναφοράς για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριο στόχος είναι να πληροφορεί αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και το κοινό και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Ο κύριος Ρουμπίκ θα μας παρουσιάσει τα απορίσματα της μελέτης επιπτώσεων όσον αφορά την αύξηση της διατροφικής παραγωγής, της ασφάλειας των τροφίμων, ορισμένων συστημάτων και τεχνολογιών γεωρικής παραγωγής με ιδιαίτερη προσοχή για, τους, για τις μικρές εκμεταλλεύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κύριε Ρουμπίκ, έχετε το λόγο όσο χρόνο χρειάζεστε μέχρι και μία μισή ώρα. Ναι, καταρχά να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Επιτροπή Ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία που μα δίνετε. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει το μιλάμε για μια δυνατότητα εξέταση των δυνατοτήτων για το μέλλον με διάφορα τεχνολογικά υπόβαθρα. Η ΣΤΟΑ, λοιπόν, ζητήσει και το 84 και δημιουργήσει και το 87 ένας ε, αντιπρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, τέσσερα μέλη της ε, Επιτροπής ΕΙΜΚΟ, Μεταφορών και το καθεξής από διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου για θητεία 2,5 ετών και φυσικά το Προεδρείο της ε, ΣΤΟΑ έχει δύο αντιπροέδρους και συμμετέχει λοιπόν και ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Η ιστορία της ΣΤΟΑ ήταν η εξής. Καταρχάς, ζητήθηκε η συνδρομή της για επικίνδυνες ε, περιπτώσεις, ε, για τομείς ε, μεγάλης επικίνδυνοτητας. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιοι τομείς στους οποίους πραγματευόμαστε στο Κοινοβούλιο, όπου θα πρέπει να λαμβάνουμε παρατάφτα τις σωστές αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια η ΣΤΟΑ μετατράπηκε, αν θέλετε, σε ένα μέσο πρόβλεψης για το μέλλον σε διάφορους τομείς. Αποφασίσαμε λοιπόν να υπάρξει συγκέντρωση σε μεγάλα project πολυετούς διάρκειας, ώστε να υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες, με... σε τομείς στους οποίους συμμετέχουν διάφορες επιτροπές, προκειμένου και οι επιτροπές να έχουν την δυνατότητα να α, συμμετέχουν. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται από ανάδοχους και οι μελέτες περιλαμβάνουν την έρευνα για την εξέβρεση των σχετικών στοιχείων που αφορούν τον εκάστοτε τομέα στην Ευρώπη. Συμμετέχουν επίσης τα πανεπιστήμια και πάντα. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η επαφή με τα πανεπιστήμια και πέρα από τα μεγάλα αυτά project έχουμε και εργαστήρια για μικρά project για το μέλλον. Κάναμε κάποια έρευνα από τον κόσμο των, της επιστήμης. Εξετάσαμε και τους, ε, την άποψη των ανάδοχων και καταλήξαμε στους τρεις τομείς που έχουμε καταλήξει. Εξετάσαμε εντελεχώς το τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες ε, τις αγροτικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπετε λοιπόν τη μελέτη που έχουμε μπροστά μας. Την, μπορείτε να την πάρετε και από την αίθουσα μπροστά. Θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε στον τομέα αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη βασική μελέτη και έξι μελέτες εν είδη προσαρτήματος, οι οποίες μας καταδεικνύουν πού θέλουμε να καταδείξουμε. Έχουμε ένα παράρτημα που α, τραγματεύεται το βρόχινο νερό και πώς μπορούμε να το συλλέξουμε. Γιατί σε πολλούς τομείς και σε πολλές περιοχές ε, ο κόσμος χαίρεται όταν βρέχει, αλλά δεν ε, έχει απαραίτητα τα μέσα που απαιτούνται για να του συλλέξει το νερό αυτό το βροχινό. Γιατί πρέπει να εγγυόμαστε και την ποιότητά του. Άρα αυτό είναι το πρώτο παράρτημα. Πώς μπορεί να γίνεται καλύτερη η συλλογή του βρόχινου νερού. Δεύτερο τμήμα, η διατήρηση της ε, γεωργίας που ασφαλώς θέτει ένα βασικό ερώτημα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Τρίτο θέμα, η πιο εντατική καλλιέργεια του ρυζιού. Γιατί φυσικά το ρύζι αποτελεί στις αναπτυσσόμενες χώρες βασική πηγή διατροφική. Ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, Ξέρετε ότι οι τιμές των τροφίμων και του νερού ακόμα αυξάνονται. Γιατί και η ανανεώσιμη ενέργεια πολλές φορές προέρχεται από τα αγροτικά προϊόντα. Άρα υπάρχει ένας νέος ανταγωνισμός μεταξύ της ε, παραγωγής ενέργειας και της παραγωγής τροφίμων. Και ξέρετε ποιε συζητήσει διεξάγονται στο Κοινοβούλιο, κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται τα δημητριακά, για παράδειγμα, για ανανεώσιμε ενέργειε. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την, αγροτική, την συγγνώμη, Επιτροπή Γεωργική ανάπτυξη αλλά και άλλε επιτροπέ. Τέταρτο παράρτημα για την ε, βιολογική καλλιέργεια. Πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε, ποιοι τομείς είναι οι πιο κατάλληλη για βιολογικές καλλιέργειες. Στο παράδειγμα 5 έχουμε τα συστήματα σοκομιάς. Ξέρουμε όλοι τι συζητήσει γίνονται για τα τροπικά δάση. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια συστήματα διατίθενται και πού μπορούμε να υποστηρίξουμε τα συστήματα αυτά. Είναι σημαντική η μελέτη αυτή για το άμεσο μέλλον, θεωρώ. Παράτημα 6. καλλιέργειες διαγωνικές. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα έντονες ε, οι συζητήσεις που γίνονται για το θέμα αυτό, transgenic crops. Και πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε και στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Γιατί λοιπόν η ΣΤΟΑ έκανε αυτή τη μελέτη, γιατί ο μισός κόσμος ζει σε αγροτικές ε, περιοχές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποσαχάρη Αφρική. Μιλάμε για ένα ποσοστό 75% που ζει στην Ήπεθρο. Στην ε, Ασία το ποσοστό αυτό είναι 50%, ενώ στη Λατινική Αμερική είναι 10% το ποσοστό αυτό. Είναι τεράστιες λοιπόν οι διαφορές που υπάρχουν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική η ενίσχυση της γεωργικής ανάπτυξης για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και την διαφοροποίηση. Άρα οι σχετικές γνώσεις και η σχετική επιστήμη σε ό,τι αφορά τι γεωργικές καλλιέργειε είναι εξαιρετικά σημαντικές και θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθηθεί η ερευνακή ανάπτυξη και στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο να μην κοιτάμε μόνο και τι γίνεται στην Ευρώπη, να δούμε ποιε είναι οι διεθνεί εξελέξει, τι σημαίνει για μα η αλλαγή του κλίματο. Πολλοί τρόποι υπάρχουν για να συνδράμουμε και στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων, για να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση τουλάχιστον. Παραδείγματα. Θεωρούμε ότι η γεωργή μικρής κλίμακας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Και θα πρέπει λοιπόν αυτοί να είναι εκείνοι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να έχουν διαφορετικές ε, δυνατότητες, να έχουν εναλλακτικές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την καλλιεργία τους, τις καλλιεργίες τους. για την διατήρηση των, ε, του εδάφους. Συνολικά λοιπόν θεωρώ ότι οι έρευνες αυτές είναι πάρα πολύ ωφέλιμες, διατίθενται όλα στο διαδίκτυο και θα χαρούμε ιδιαίτερα αν οι αντιπροσωπείες από τις αναπτυσσόμενες χώρες λάβουν και τις ε, μελέτες της ΣΤΟΑ πέρα από τις υπόλοιπες πληροφορίες που λαμβάνουν. Αυτό θεωρώ ότι θα βοηθούσε ιδιαίτερα στον τομέα αυτό. Κλείνοντας, να αναφέρω κάποια μεγάλα project που έχουμε για, το, για τα επόμενα τρία έτη. Ένα συγκεκριμένο project, το οποίο και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. οικολογικές και αποδοτικές μεταφορές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ υψηλή προτεραιότητα. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε και τον κόσμο και τα προϊόντα από και προς τις μεγάλες πόλεις. Σημαντικό θέμα. Κατά δεύτερον, βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση μάλλον των ε, ανανεώσιμων πόρων. Ενέργεια, νερό. Έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις και θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Και τρίτο θέμα, είναι η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα κοινωνικά δίκτυα και πώς μπορούν αυτά να βοηθήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και καλύτερη ανταπόκριση. Επίσης, οι δυνατότητες ε, εκπαίδευσης μέσω κοινωνικών δικτύων, κατά πόσον είναι σωστός, το σωστό μέσο εκπαίδευσης κτλ. Σας παρουσίασα λοιπόν αυτά τα σημεία, ωστόσο να, θα χαρώ να μου κάνετε και ερωτήσει. Ευχαριστώ, κυρία Κέλλερ. Yeah, your... Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, πώς θα γίνει η κατανομή των αποτελεσμάτων και γενικά η δημοσιοποίησή τους μέσω του website, είπατε. Είπατε ότι θα τα, θα δημοσιοποιήσετε, αλλά θα γίνει πως και με άλλους τρόπους. Πώς θα διαδοθούν αυτές οι πληροφορίες, γιατί είναι πολύτιμα τα στοιχεία που θα έχετε. Κάτι άλλο επίσης, δεν ξέρω αν φαίνομαι άσχετη, αλλά πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ποιος αποφασίζει τι θα κάνετε. Άμα εμείς κατεβάσουμε μια ιδέα, τι θα κάνουμε, θα σας βρούμε. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ο Ρούμπι είχε, είχε να μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το πώς έχουν τα πράγματα και τι γίνεται με το ΣΤΟΑ και το πάνελ του ΣΤΟΑ. Τι είναι με τι αναπτυσσόμενες χώρες, πράγματα τα οποία εδώ δεν τα ξέρουμε γιατί στην Αφρική αλλά και στην Ασία δεν υπάρχουν τράπεζε και κανονικοί λογαριασμοί και προσπαθούν να αντικαταστήσουν τράπεζες με κινητά τηλέφωνα. Και σε μακρινά σημεία της Αφρικής. Δεν υπάρχουν αυτό μηχανές, ε, υποκαταστήματα τραπεζών και τέτοια. Και γι' αυτό έχει ε, υπάρξει ανάγκη για όθηση στην τεχνολογία που θα τους βοηθήσει. Άρα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, να εισαγάγουμε τη σχετική τεχνολογία και στην Ευρώπη. Να γίνει μια σχετική μελέτη ενδεχομένω γιατί είναι εκατομμύρια εκείνοι που πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων στην Αφρική Νοτιού Σαχάρας. Δεύτερο σημείο κύριε Βίλη. Ξεκίνησα και εγώ ένα project για διανομή φορητών υπολογιστών και έχουμε φτάσει τώρα στα 27 εκατομμύρια. Φτάσαμε μέχρι και την Παπούα. Μιλάμε για κόσμο που δεν έχει καν ηλεκτρισμό και τα φορτίζουν με την ενέργεια του ηλίου. Τέτοια, τέτοιους φορτούς υπολογιστέ προωθήσαμε. Το χρησιμοποιούν τα παιδιά στα σχολεία για να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Άρα για αυτούς είναι τεχνολογικό άλμα Μιλάμε για μέρη που δεν έχουν ούτε δρόμους. Και πριν από κάνα δύο αιώνε ζούσαν σε συνθήκε πρωτόγονες. Έχουν τώρα επομένω φορητούς υπολογιστέ. και μιλάμε για σχολεία που δεν έχουν ηλεκτρικό. Όμως έχουν διαδίκτυο και επικοινωνούν έτσι. Πρόκειται για άλματα καθώ προχωρεί η τεχνολογία και επομένω είναι τεράστιε αυτέ οι ευκαιρίε για χώρε, χώρες ώστε να υπερβούν τα πρώτερα στάδια της εκβιομηχάνησης. Έχουν δηλαδή κοινέ πληροφορίε, δεν έχουν εργοστάσια, αλλά έχουν την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας επομένως. Λάβετε τα αυτά υπόψη, να δούμε πώς μπορούμε για τα αντισιακά μας προγραμματα όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε. θα λάβω τώρα τον λόγο για να σας ερωτήσω κύριε Ρουμπίχη, πώς θα εξασφαλίσετε ούτω ώστε οι μελέτες και αυτές οι γνωμοδοτήσεις είναι επιλαγμένες από την επίδραση των λόμπι Φερρυπίν αφορά αυτές τις γενετικές τροποποίησεις. Υπάρχει διάφανη λειτουργία ούτω ώστε να ξέρετε ε, μήπως επηρεάζεται κατά αυτόν τον τρόπο κάποιος από τους επιστήμονες που σας βοηθούν. Δεν ξέρω τώρα μήπως θέλει να λάβει τον λόγο η Κομισιόν και κατόπιν θα ξαναλάβει τον λόγο για να δευτερολογήσει ο κύριος Ρίμπιχ. Όχι, δεν θέλει τον λόγο. Ούτε η Κομισιόν. Α, η Κομισιόν, ναι, ναι. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση όσον αφορά αυτές τις ε, επιλογές μειωμένης έντασης. Έχουμε και επιστροφές πάνω στο θέμα της ε, ασφάλειας των ειδών διατροφής. Για κάποια μέτρα βιώσιμης υφής και έντασης. Η δική μας ερώτηση είναι η εξής. Γιατί καταλήξαμε σε αυτές τις πέντε μελέτες, αυτές τις πέντε περιπτώσεις, αυτές τις μελέτες υποθέσεων και βέβαια προσθέσει ενδιαφέρον η υπόθεση των γενετικών μεταλλαγμένων. Όμως, μπορεί κανείς να κάνει πολλά περισσότερα όσον αφορά την παραδοσιακή τεχνολογία πολλαπλασιασμού των ειδών. Γιατί σου διαλέξετε αυτές τις ε, πέντε υποθέσεις εργασίας για Έχετε το λόγο. La parole pour la, les réponses. Yes, uh, first of all, the question of Mrs. Keller. Uh, of course, we try... Πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε και να κάνουμε γνωστές τις μελέτες μας. Ε, τις δημοσιεύουμε και στην ιστοσελίδα Κάνουμε πολλές συναντήσεις και εργαστήρια και με τους ειδικού τους εμπειρογνώμονες και έτσι καθίσταται σαφές ότι δεν είμαστε μονόπλευροι. Όπως και στο Κοινοβούλιο, όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και για το κοινό, αν ενδιαφέρεται. Για να ακούγονται και διάφορες γνώμες. Από την άλλη, τα αποτελέσματα πάντα παρουσιάζονται και στις συνεντεύξεις τύπου, κατά τις οποίες προσπαθούμε να παρουσιάζουμε με δομημένο τρόπο τα αποτελέσματα, αλλά από ό,τι ξέρετε στον τομέα τον επιστημονικό χρειάζεται και ειδικού ε, δημοσιογράφους. Επιστήμονες δημοσιογράφους. Και σήμερα, για παράδειγμα, θα μπορούσα να βρίσκομαι στο Λονδίνο με, για να κάνω σχετικές ε, συναντήσεις, αλλά έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Και σε συνεδριάσεις του STS, η επιστημονική κοινότητα έδειξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ερευνών της ΣΤΟΑ. Δεύτερη ερώτηση ήταν πώς η... γίνεται η λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό της ΤΟΑ. Φυσικά, καταρχάς, υπάρχει το Προεδρείο. Υπάρχει επίσης και το πάνελ. Συνερχόμεθα λοιπόν. Το project ε, για το 2010 αποτέλεσε έτοιμα της επιστημονικής κοινότητας. Είχαν τεθεί πολλές ιδέες, αλλά συζητήθηκαν λοιπόν όλες αυτές οι ιδέες από τις πολιτικές ε, επιτροπές και από τις επιστημονικές ε, ομάδες και οι αποφάσεις, ε, η απόφαση που λήφθηκε για την επιλογή των προγραμμάτων λήφθηκε με ομοφωνία από όλες τις πολιτικές ομάδες. Για τον κύριο Ντέβα, φυσικά η κινητή επικοινωνία και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ε, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όλο ένα και αυξανόμενο ρόλο και μιλάμε για κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ. Και στους τομείς αυτούς Ε, μάλλον τους τομείς αυτούς τους εξετάζουμε και στον μεγάλο κλάδο των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γιατί στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να διασφαλίζονται τα συστήματα πληρωμών για να είναι σίγουρα. Χρειάζεται λοιπόν ταυτοποίηση από τον καταναλωτή, αλλά και από την άλλη πλευρά, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή ποιος επικοινώνησε με ποιον, για να μην ανακυπτούν σφάλματα. Στο μέλλον, από ό,τι ξέρετε, θα υπάρχουν πολλές πιο πολλές δυνατότητες και μέσω των κινητών τηλεφώνων. Αναπτύσσεται λοιπόν γοργά η τεχνολογία και είναι σημαντικό να επιμείνουμε στον τομέα της ασφάλειας. Επικεντρώνεται λοιπόν η ΣΤΟΑ στην πτυχή αυτή της ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οπουδήποτε δηλαδή χρειάζεται αμφίδρομη επικοινωνία και ταυτοποίηση. Η Πρόεδρος ρώτησε πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λόμπι δεν θα ασκήσουν υπερβολικά μεγάλη επιρροή. Καταρχάς, πρώτη ασφαλιστική δικλίδα είναι το Κοινοβούλιο, γιατί ξέρετε ότι συμμετέχουν πολλές χώρες, πολλές πολιτικές ομάδες, είναι πολλά και διάφορα τα συμφέροντα που υπάρχουν στην Επιτροπή μας. Και στο επίπεδο αυτό έχουμε και ανεξάρτητους ε, συμβούλους οι οποίοι επιλέγονται από την διάσκεψη των Προέδρων για τριετή θετία, άρα δεν τους επιλέγουμε εμείς, τους επιλέγει η διάσκεψη των Προέδρων. Και φυσικά έχουμε και εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για όλους τους διάφορους τομείς. Αυτό που είναι καινούριο και αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε για τα μεγάλα project είναι να υπάρχει ε, έλεγχος από αμοτήμους, διακή παρακολούθηση και έχουμε και άλλες ε, δραστηριότητες υπόψη μας για τη βελτίωση της, ε, του ελέγχου από αμοτίμους αυτό που ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί επιλέξαμε τους διάφορους τομείς για να κάνουμε τις μελέτες. Ήταν οι τομείς που μας αναφέρθηκαν. Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε αυτά τα κρίσιμα σημεία. Να αναζητήσουμε τεχνολογικές λύσεις σε τομείς οι οποίοι συζητιούνται έντονα σήμερα. Είδαμε λοιπόν πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτά τα θέματα. Και φυσικά, αν διαβάσετε τις μελέτες αυτές, θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας και θα θέλαμε και μια, τελευταία, μια επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Κατά τελευταίο σας προσκαλούμε κάθε πέμπτη στις 9.30 συναντιόμαστε στο Στρασβούργο επί μία μισή ώρα. Ναι, είναι ένα πρωινό γεύμα. Ναι, από ό,τι ξέρετε βέβαια δεν έχουμε κρουασάν, έχουμε μόνο καφέ και τσάι. Αλλά γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αν υπομονούμε να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας πληροφορίες. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να έρθω να σας αναφέρω τα επιστημονικά αποτελέσματα της επιστημονικής αυτής ε, εργασίας που γίνεται. I just opened your study uh, transgenic crops. Μόλις είδα τη μελέτη για τα transgenic crops, για τις uh, καλλιέργειες transgenic, υπερφυτά transgenic για την καταπολέμηση της υποσυτισμού, μια από τις προκλήσεις σε θέματα υγείας. αλλά δεν φαίνεται καν να το συζητήσετε το θέμα αυτό. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό δεν ελυθεύει ως πρόταση. Να δώσουμε δηλαδή τρόφιμα για όλο τον κόσμο, να εξασφαλίσουμε τρόφιμα χωρίς τέτοιου είδους φυτά που ξεπερνάνε το ένα είδος. Στη σελίδα 21 βλέπω ότι είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά τα θέματα της παγκόσμιας υγείας. If before Mr. Rubik answers that question. Πριν απαντήσει ο κύριος Ρούμπικ, λέει ο κύριος Ντέβα, θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση σχετική θα πεινούσε σήμερα ο κόσμος, ιδιαίτερα στην Ινδία, θα ήταν ο μισός ο πληθυσμός της Ινδίας, αν δεν υπήρχε μια νέα καλλιέργεια που δημιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 80 από ένα δανό καθηγητή, ο οποίος ε, μετασχημάτισε τον κόσμο και έσωσε δισεκατομμύρια ζωές. Διαγωνιδιακή καλλιέργεια ήταν κι αυτή και έθρεψε τον κόσμο. έσωσε δισεκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, εγώ δεν θα ανησυχούσα και πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος απλώς επισήμενα ότι το θέμα αυτό συζητιέται. Και ο κύριος Ρουμπίκ, όπως ξέρετε, μελέτες του 2008, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, έγινε αυτή η μελέτη και φυσικά η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ημερήσια διάταξη και η Κομισιόν κάτι έκανε σχετικά. Τα κρατημέλη, η Κομισιόν, οι επιστήμονες, δεν υπάρχει λύση 100%. Η γεωργία είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Το παγκόσμιο εμπόριο, υπάρχουν πολλά συμφέροντα, δεν είναι μόνο τεχνολογικές λύσεις. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές που αφορούν τον τομέα αυτό. Εμείς κοιτάμε, οι μελέτες μας δεν είναι κοντά στην τεχνολογία και όχι κοντά στις πολιτικές αποφάσεις. Εμείς να, θέλουμε να τονίσουμε τι ευκαιρίες υπάρχουν και οι πολιτικοί θα αποφασίσουν ποιο μοντέλο ταιριάζει για κάθε χώρα, για κάθε αναπτυσσόμενη χώρα. Γιατί και οι χώρες αυτές μεταξύ τους έχουν διαφορετικές δομές και διαφορετικά προβλήματα και δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Εμείς παρουσιάζουμε τις διάφορες λύσεις που υπάρχουν έτσι ώστε οι πολιτικοί να επιλέξουν. Πρόεδρος. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Μελέτη μια πρόταση ψηφίσματος από δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν σχετικά με την ε, Σύνοδο Κορυφής Αφρικής Ένωση. Οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια πρόταση ψηφίσματος πριν τη διάσκεψη αυτή υπήρξε ετοιμα να ανακληθεί αυτή η απόφαση με νέα συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο θα γίνει αυτό, αλλά η συζήτηση θα γίνει σήμερα. Η τρίτη διάσκεψη κορυφής Ένωση θα γίνει στη Λιβύη 29 και 30 Νοεμβρίου με συμμετοχή του Πρόεδρου Μπούζεκ. Με την προσωπία του Κοινοβουλίου θα περιμένουμε σε μια προδιάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο, όπου οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και του Πανεφρικανικού Κοινοβουλίου θα εγκρίνουν μια κοινή δήλωση για τη στρατηγική που θα μπει ως παράδειγμα στα πορίσματα της διάσκεψης κορυφής. Η δεύτερη διάσκεψη κορυφής το 2007 πρόθεσε μια φιλόδοξη στρατηγική συνεργασία των δύο υπήρων και για την ανάπτυξη και για πολλούς άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Τα τρία χρόνια που πέρασαν, η αρχιτεκτονική αυτή της στρατηγικής άρχισε να εφαρμόζεται. Δώσαμε μάχη ώστε στην κοινοβουλευτική διάσταση να λαμβάνεται παρκώς υπόψη στον πολιτικό διάλογο και στην εφαρμογή των πρωτοβουλειών. Από τη διάσκεψη κορυφής περιμένουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης που ελπίζουμε να δώσει συγκεκριμένα πορίσματα πέραν των εργασιών που γίνονται για τις ε, θεσμικές δομές. Στη, το Νοέμβριο θα υπάρξει μια δήλωση στην ε, Ολομέλεια εκ μέρους Κομισιόν και του Συμβουλίου. Όλοι έχετε πάρει ένα σχέδιο του ψηφίσματος που θα εγκρίνει το Νοέμβριο πριν τη διάσκεψη κορυφή στο Κοινοβούλιο προς γνώση των Πρωθυπουργών στην Τρίπολη. Είμαι η συγγήτρια του ψηφίσματος αυτού στο όνομα της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πριν δώσω το λόγο στους βουλευτές μας, θα ήθελα να ακούσουμε τον Μάικελ Γκάλερ, που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος, κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο όσο χρόνο χρειάζεστε. Γιατί σήμερα ειδικά δεν βιαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω εδώ. Είναι λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστώ που ξαναβρίσκομαι στην παλιά μου κοινωνική επιτροπή και βλέπω όλους αυτούς τους ε, παλιούς γνωστούς και συνάδελφοι ακριβώς όπως προείπε η πρόεδρος έτσι έχει η διαδικασία θα έχουμε την προπαρασκευαστική συνάντηση το απόγευμα της 27ης ενδεκάτου μέχρι τώρα. Ακολουθεί τη διαδικασία που αποφασίστηκε στην Λισαβόνα προτριετία. Και από κάθε πλευρά έχουμε 25 μέλη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο στη δεύτερη συνάντηση κορυφή δόθηκε καινούργια όθηση αυτή τη ε, κοινή στρατηγική που την επεξεργαστήκαμε τότε και τώρα ήρθε η ώρα να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Στο Μαλάβι κανονικά θα γινόταν αυτή η συνάντηση, γιατί αυτοί έχουν την Προεδρία, όμως δεν έχουν απαραίτητη υποδομή και έτσι η προηγουμένη Προεδρία προσφέρθηκε να διοργανώσει και την φετινή συνάντηση. Πρώτη αυθορμήτως συγκροτήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία η αντιπροσωπεία και είχε προβλεφθεί μια μακρότερη περίοδος και είπαμε αυτό δεν θα κρατούσε μόνο για μία συνάντηση οπότε το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτή την στατική στην υλοποίησή τη. Μόνιμη αντιπροσωπή επομένω, όπως τότε και οι συνάδελφοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και όπως ε, γνωρίζετε αυτό το οποίο θέλουμε τώρα είναι να υπάρξει μια κοινή θέση. Να, προ 15 ημέρου συντάξαμε αυτό το κείμενο, αυτό το σχέδιο κειμένου της δήλωσης. Δεν ξέρω αν το έχουν λάβει όλοι. Καλά, θα σας το δώσουν. στην Τρίπολη πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό. Θα λάβει το χαρακτήρα και το ύφος μιας δήλωσης, το σχέδιο κειμένου και τη Δευτέρα θα φύγουμε για την συνάντηση της Κινσάσα. Οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου και του Πανεφρικανικού Κοινοβουλίου επίσης πρόκειται να συναντηθούν στην Τρίπολη και επαναλαμβάνω ότι αυτό το γύρο πέρασε, καταλήξαμε κάποιες κοινέ θέσεις. Πρώτα-πρώτα, έχουμε εμπλακεί σε αυτές τις υπουργικέ ε, τριμερείς συναντήσεις και το κάναμε σαν εξαμερή διάλογο Και αυτό καθιερώθηκε να προηγείται τη υπουργική συνάντηση, ούτω ώστε να συζητούνται ε, οι απόψει των κοινοβουλίων όσον αφορά την υλοποίηση των προτάσεων για την κοινή στρατηγική. Αυτό βέβαια δεν απέδωσε πάντα, παρά το ότι η καταρχήν συμφωνία. Κάποιες κυβερνήσεις από αφγανικής πλευράς προσπάθησαν να γνωρίσουν τα συμπεφωνημένα. Εμείς όμως χτυπήσαμε κατά κάποιο τρόπο το χέρι στο τραπέζι για να τους ε, υπενθυμίσουμε ότι δεν μπορούν να αγνοούν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί όσον αφορά τα κοινοβούλια και το ρόλο τους. Είναι πολύ σημαντικά τα κοινοβούλια για την στρατηγική αυτή. Αυτό τώρα το οποίο διαπιστώθηκε είναι ότι γενικώ υπήρξαν επικρίσεις για την έλλειψη δέσμευσης πολιτικής αποφασιστικότητας για την υλοποίηση στρατηγικής αυτής. Και επίσης επικρίθηκε και το ότι η πολιτική συνάντηση δεν ήταν ουσιαστικά υπουργική. Συνάντηση, συνεδρίαση ήταν ουσιαστικά δίπλα εργασίας. Όμως βέβαια θεωρούν οι Αφρικανοί συνομιλητές μας ότι τους σεβόμεθα και ότι λαμβάνεται όπως το λένε και εμείς επιμείναμε στο ότι θα πρέπει να προσδίδεται η απαραίτητη σημασία σε αυτές τις συναντήσεις. Είναι κάπως περιπλοκή δομή, έχουμε τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων, έχουμε την, αυτή την υπουργική τρόικα, έχουμε κάποιες άλλες συναντήσεις. Α, ναι, και είναι και διάφορες task force. Άρα έχουμε τις ε, expert groups των εμπειρογνωμόνων, έχουμε τα task groups, μετά έχουμε τις τρόικες των υπουργών, αλλά η πολιτική καθοδήγηση του ΣΥΠΗΝ δεν υπάρχει. Ο καθένας είναι ειδικό στα θέματα του, έχει τις προτάσεις του, όμως εάν δεν υπάρξει πολιτική δέσμευση, αποφασιστικότητα και κατευθυντήρια γραμμή, δεν θα έχουν αποτελέσματα. Γιατί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα και αυτή θα είναι προστιθέμενη αξία για την συνεργασία Ένωσης και Αφρικής. Είχαμε πει ότι κάτι θα γίνεται από τρία χρόνια, περάσανε. Τι έγινε. Θα είχε γίνει τίποτα αν δεν υπήρχε αυτή η στρατηγική, αν είχαμε μείνει στη φάση της Κοτονού, στις παλαιότερες μορφές δηλαδή συνεργασίας, αν δεν είχαμε αυτή την κοινή διάσκεψη. Άρα αυτό ανεστούμε τώρα ε, κάπως να προκύψει είναι αξία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τάξουμε και τις προτεραιότητες. Και δεν μπορεί να έχει κανείς πολλές προτεραιότητες. Λέγεται ότι έχουν οριστεί 22 θέματα προτεραιότητας. Δεν είναι και τόσα πολλά. και γι' αυτό καταλήξαμε στο συμπέρασμα οι συγκεκριμένες προτεραιότητες να είναι πιο λίγες και βέβαια θα πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να προτείνουν και οι Αφρικανοί συνάδελφοι. Βασικό τους θέμα είναι η διατροφική ασφάλεια, κορυφαία τους προτεραιότητα. έχει γίνει μείωση των κονδυλίων που διαθέτουν ε, τα κράτη της Αφρικής για την υπόθεση αυτή, από 20% στο περίπου, η μείωση. Και ανέβηκε η τιμή των τροφίμων και να ξέρετε ότι αυτοί που επενδύουν στην Αφρική για παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιούν την Αφρική τη γη τη, αλλά παράγουν για τον εαυτό τους. Επομένως, είπαμε ότι στις προτεραιότητες δεν αρκεί να η διδροφική ασφάλεια να είναι μια υποπαράγραφος, ένα υποσημείο θα πρέπει να είναι ένα αυτόνομο σημείο. Μόνο του πρέπει να είναι στην μέση διάδειξη του ΣΥΠΗΝ. Για τα θέματα ασφάλειας πάει καλά η συνεργασία. Αυτό δεν εκπλήσει βέβαια, γιατί όταν έχουμε κάποια συγκρούσει τα πράγματα είναι κατεπίγοντα, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα, θα πρέπει κανένα να αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά. Οπότε, εκτό από το θέμα τη ειρήνη για την Αφρική, πρέπει να αποφασίζει ποιε δραστηριότητε υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα λοιπόν αυτό και βοηθάει. Και γι' αυτό και σε αυτό το μέτωπο πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα, εν ώψη της συνέντευξης κορυφής, ζητήθηκε να δούμε τι, αν έχει κυρωθεί αυτός ο χάρτης για τα βασικά εκλογικά και συναφή δικαιώματα. Αυτό έχει τη μορφή της συμφωνίας, αλλά αν δεν το έχουν κυρώσει αυτό το κείμενο αρκετά κράτη, πότε θα δρανοποιηθεί. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς ε, συναδέλφους να προβάλλουν το θέμα αυτό, να υπάρξει αυτή η προβολή παντού, εργαστήρια και τέτοια. Προσπογράφηκε λοιπόν αυτό το κείμενο, αλλά πρέπει να κυρωθεί, θα είναι κρίμα αφορά δημοκρατία, διακυβέρνηση, εκλογές. Θα είναι κρίμα επομένως αυτό το κείμενο να αδρανοποιηθεί ελήψη υποστήριξη. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά την διαδικασία. Μου είπαν η διάσκεψη των Προέδρων ήδη αποφάσισε, όπως είπες Πρόεδρε, να συζητήσει πριν γίνει η συνάντηση κορυφή, τα σχετικά και τον Δεκέμβριο ίσως να προωθηθεί ένα ψήφισμα για το αποτελέσμα. Όσον αφορά τώρα την αντιπροσωπεία, κατεπηγόντως, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπροσωπεία εκτός προσώστοσης, να μην χρησιμοποιηθεί επομένω η ποσότητα που αφορά αντιπροσωπείε, κοινοβουλευτικέ και επιτροπέ, γιατί είναι εδώ κάτι το έκτακτο, είπαμε. Η εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε τριετία. Είχαμε 25 τελευταία φορά, αλλά από ό,τι μου λένε, και αυτό ακόμα μπορεί να διορθωθεί, εάν δεν έχουμε ένα άνετο νούμερο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δώδεκα συν τρεις είπαμε. Εσύ πρόεδρε, ο Λουιμισελ, ο Μπούζεκ και άλλοι δώδεκα δηλαδή από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Και όταν μπορέσουμε να βρούμε τους 12, συν τους άλλους τρεις, θα είμαι ευχαριστημένος, αλλά να δούμε. Ο κανόνα συνεχίζει να ισχύει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η ποσόστοση, αλλά αυτό κάπως με δυσκολεύει και από πολιτική πλευρά. Θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι αποφάσει που θα προκύψουν. Θα πρέπει να είμαστε παρόντε και όχι απόντε στη λήψη των αποφάσεων να γίνει αυτό όπως πρέπει. Και η προσοχή είναι αυτή που πρέπει. Έχουμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Εγώ έχω να πω ότι στο, για το σημείο 6... Εδώ υπάρχει ένα θέμα πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τα, τα δύο σώματα τα οποία έχουν προβλεφθεί. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι επειδή υπάρχουν δυσκολίες από των Αφρικανικών Κοινοβουλίων όσον αφορά τη συνεργασία μας μαζί τους. Είπαμε πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δυνατότητες αυτές που δεν έχουν. Και έτσι να μπορούν τα κοινοβουλία αυτά να ασκούν τον κοινοβουλευτικό δημοκρατικό έλεγχο στα πλαίσια του συντάγματος της χώρας τους. Είπαμε για την υλοποίηση της στρατηγικής, αυτό δεν αρκεί όμως. Θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη αρμοδιότητα και κυρίως γιατί ε, αν τους δοθεί η δυνατότητα θα κάνουν αυτό που συνταγματικά προβλέπεται να ασκούν δηλαδή κριτική στην κυβέρνηση της χώρας. Το οποίο είναι το σωστό και όχι εμείς να ασκούμε την κριτική αντί για αυτούς. Και επομένως είπαμε ότι η Επιτροπή θα εξοφηθεί ακριβώς το να αφουγκράζεται περισσότερο τη φωνή των κοινοβουλίων. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτε άλλο. Ε, Ευχαριστώ να απαντήσω. Κύριε Ντίβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή ο κύριος Γκαλρέ είναι πολύ ενημερωμένο σε τέτοια θέματα, ε, γενικότερα και σε ό,τι αφορά την ε, Αφρική, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, διάφορες δομές που έχουν δημιουργηθεί για να επιτύχει η Σύνοδος ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Να θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα στον κύριο Γκάλερ, το οποίο με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην παράταση των Εθνικών Κοινοβουλίων όμως. Και στα Εθνικά λοιπόν Κοινοβούλια. Οι εκλεγμένοι πρέπει να είναι υπόλογοι και πώς είναι υπόλογοι απαντούν στις ερωτήσεις των κοινοβουλίων. Για παράδειγμα, έρχεται ο, Ευρωπα... ο κ. Μπαρόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απαντάει σε ερωτήσεις. Πόσα αφρικανικά κοινοβούλια έχουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο πρόεδρος των Αφρικανικών κρατών, για παράδειγμα, πηγαίνει στο κοινοβούλιο ή απαντά μέσω του Πρωθυπουργού του ε, σε τέτοιες ερωτήσεις. Είναι υπόλογος για όσα κάνει. Γιατί αν μπορούμε να εισάγουμε την διαδικασία αυτή και αν μπορούμε να δώσουμε τέτοια δύναμη στα μέλη του Κοινοβουλίου στην Αφρική προκειμένου να εκτελούν την εξουσία τους χωρίς να φοβούνται ότι θα μπουν στη φυλακή την επόμενη μέρα επειδή έθεσαν ένα ερώτημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, ασυλία και την δυνατότητα τέτοιας υποβολής ερωτημάτων. Αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της καλύτερης διακυβέρνησης στην Αφρική. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο θεωρούμε αυτονόητο, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν είναι εγγυημένη αυτή η δυνατότητα, ε, δεν θα κάναμε τίποτα. Και ρωτώ λοιπόν το μας. αυτό υπάρχει, αυτό δυνατότητα, απάντηση. Οι χώρες που έχουν το βρετανικό σύστημα τουλάχιστον, στο, στη θεωρία έχουν τέτοια πρόβλεψη. Ε, ειλικρινά να σας πω, πρέπει να ομολογήσω, δεν ξέρω κατά πόσον χρησιμοποιείται και εφαρμόζονται καταλήλως το σύστημα αυτό. Αλλά ξέρω για παράδειγμα ότι στην κυβέρνηση της Νοτιού Αφρικής θέτουν τέτοια ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι απαραίτητα ο πρόεδρος εκείνος που απαντά. Στα άλλα κοινοβούλια, στην Αμίμπια, επίσης τίθενται ερωτήματα και σε ό,τι αφορά την γαλλόφωνη Αφρική, στο κοινοβούλιο του Μάλι, για παράδειγμα, ξέρω ότι ακόμα και δύσκολα ερωτήματα ε, τίθενται. Και νομίζω λοιπόν ότι και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό. Είμαι βέβαιος και είμαι πεπισμένος ότι γίνεται αυτό. Αλλά για να αντιστρέψω την κατάσταση, ξέρουμε τι μπορούμε να ρωτήσουμε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Και ξέρουμε πόσο πόσο είναι και οι απαντήσεις και ακόμα και αν το ξέρουμε ότι συνήθω είναι, υπεκφεύγουν ε, στι απαντήσεις τους, προσπαθούμε να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και παρόλα αυτά καταφέρνουν να υπεκφεύγουν. Αυτή λοιπόν η ενίσχυση των ε, βουλευτών θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη υποβολή των σωστών νομοθετημάτων, αλλά θα πρέπει φυσικά να είναι σε θέση να καταθέσουν τον προπολογισμό, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. για να μην προέρχονται όλες οι νομοθεσίες από το εκτελεστικό σκέλος της εξουσίας, να συμμετέχει και το κοινοβουλίο. Αυτό σπάνια χρησιμοποιείται. Υπάρχει ω θεωρητική δυνατότητα, αλλά δεν αξιοποιείται. Και αυτό θα αποτελούσε ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τους βουλευτές και το προσωπικό τους για την κατάρτιση νομοθεσίας. Θα μπορούσε να καταρτιστεί ένα σχετικό πρόγραμμα για τα κοινοβούλια σε ό,τι αφορά, αφορά δηλαδή κατάρτιση προπολογισμού, νομοθεσίας, υποβολή των ερωτημάτων. σε ό,τι αφορά δηλαδή τα πολιτικά θέματα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ορισμό της εργασίας ενός βουλευτή και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο υπάρχουν επίσης, ε, υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων. Και συμμετέχουν και οι επίτροποι, αν και δεν συμμετέχουν ε, πάρα πολύ καλύπτουν, αν θέλετε, ε, καλύπτουν λίγοι πολλά θέματα. Και αυτό συμβαίνει και στο Στρασβούργο. Πολλέ φορέ ένα επίτροπο απαντά για θέματα άλλων συναδέλφων. Ναι, έχουμε ακόμα δύο μιλητέ. Θα απαντήσετε στο τέλο. Ο κύριο Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα. Να μιλήσω μήπως τα Ολλανδικά. Για να είμαστε πιο απλοί. για να ξεκουραστεί η καμπίνα. Να αναφέρω κάποια στοιχεία. Η Σύνοδος Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όταν θα γίνει θα ήθελα ε, να θέσουν και κάποια θέματα. Θεωρούμε στην ομάδα μας ότι η στρατηγική για την Αφρική είναι πάρα πολύ όμορφα διατυπωμένη στην στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά ενώ ναι, η διατύπωση είναι πάρα πολύ ωραία, Τώρα θα πρέπει πλέον να φροντίσουμε να δοθεί μια νέα όθηση στην στρατηγική αυτή. Και διαπιστώνουμε ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής δεν είναι τόσο ισχυρός όσο θα θέλαμε, όσο απαιτείται. Και θα πρέπει να, ε, μάλλον χρειάζεται έντονη προσπάθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την Ουγγάντα και τη στάση της απέναντι στα άτομα με διάφορε σεξουαλικό προσανατολισμό. Και επίση βλέπουμε ότι η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και από τα αφρικανικά κράτη τα ίδια, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά αναφέρονται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Θα πρέπει όμως να εφαρμοστούν καλύτερα και κάποια άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικότερα και πιο ειδικά αν θέλετε μετά την σύνοδο της Λισαβόνα πριν από κάποια χρόνια η Αφρική έχει μπει σε μια γρήγορη ε, πορεία ανάπτυξη της οικονομίας μας. Αυτό της οικονομία της. Είναι πολύ ευπρόσδεκτο αυτό, αλλά πολύ ανισομερής είναι αυτή η ανάπτυξη και η ευμερία η οποία έχει προκύψει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ευημερία. Ο πλούτος, ο οποίος προέρχεται από τις πρώτες ύλες, από το φυσικό πλούτο, γιατί σε φυσικό πλούτο οφείλεται κατά βάση, να διανεμηθεί πιο σωστά. Και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τη Σύνοδο. Να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί, να γίνουν επενδύσεις ε, στην ε, ε, υγεία, στην εκπαίδευση, στην καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, στην προστασία του περιβάλλοντο και φυσικά σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία. Τρίτο στοιχείο. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικής θα πρέπει να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Τέταρτο σημείο. Στην ε, εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική θα πρέπει να συμμετάσχουν και μη κρατικοί φορείς, προκειμένου και αυτοί να συμμετάσχουν σε ό,τι αφορά τη συνεργασία αυτή. Και το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για τα Εθνικά Κοινοβούλια και φυσικά για το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Πέμπτο στοιχείο. Η ενίσχυση της Αφρικανικής Ένωσης αποτελεί στρατηγικό στόχο, όχι μόνο για την, Ευρωπαϊκή, για την Αφρική, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η Αφρικανική Ένωση να είναι σε θέση και να έχει και τις δυνατότητες, την ισχύ, προκειμένου να δρά και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Αυτό πολλές φορές θα σήμαινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην άκρη, αν θέλετε. Αποφασίστηκε η επένδυση πόρων για την ενίσχυση της Αφρικανικής Ένωσης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το διαχειριστικό σκέλος της Αφρικανικής, ε, το επιχειρησιακό σκέλος της Αφρικανικής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει έντονη συνεργασία μεταξύ Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει, όπως αναφέρεται και στην συνθήκη της Λισαβόνας, να υπάρχει ε, συνοχή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ε, ως προς την Αφρική και δεν θα πρέπει να είναι αντίθετη η στόχη της ε, ανάπτυξης με τους στόχους του εμπορίου. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, η κυρία Κέλλερ. Thank you. I with the focus on land grabbing. Ευχαριστώ με όλα όσοι με τον πλούτο και τα άλλα υπέρ των κοινοβουλίων. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που ανεφέρθηκε για την πολιτική συνοχής. Έχουμε δεσμευτεί οι πολιτικέ μας να μην κάνουν ζημιά στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να την υποστηρίζουν. Αυτό δεν συμβαίνει και πολύ. Δεν συζητιέται πολύ. η Κομισιόν θα έπρεπε να φροντίζει και άλλες πολιτικές να είναι φιλικές ως προς την ανάπτυξη, να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, όχι να την επιζημιώνουν. Θα έπρεπε και εμείς το ψήφισμά μας να το επισημάνουμε αυτό. Επίσης, η δέσμευση να έχουμε πιο περιφερειακή προσέγγιση. Όχι με διαφορετικέ σχέσει με μία χώρα, διαφορετικέ σχέσει με τη γειτονική χώρα, μία πιο περιφερειακή προσέγγιση. Έτσι ώστε να συνεργάζονται οι χώρε με του γειτονέ του. Ελπίζω και αυτό να μπορέσουμε να το βάλουμε στο ψήφισμα. Και πριν την κορυφή αυτό, γιατί μετά, ωραία λόγια, αλλά μετά δεν επηρεάζουμε τα πράγματα. Και ελπίζω όλα αυτά να συζητηθούν και στην κοινοβουλευτική συνάντηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και η Κομισιόν, ο κύριος Καρλ Χαλ και ο κύριος Φρανσίς Τράκη. κάποια παρανόηση. Ο κύριος Τζίντζιος θα απαντήσει εξ ονόματος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σχολιάζουμε μερικά από τα σημεία που αναφέρατε. Από τη δική μας σκοπιά θεωρούμε θετική τη δράση και του Ευρωκοινοβουλίου και των Αφρικανικών Κοινοβουλίων στην κοινή στρατηγική και θα θέλαμε αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Είχαμε προπαρασκευαστικές συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα στην Αντισαμπέμπα. Κρίμα που δεν είχαμε κανένα από τα κοινοβούλια, ούτε από την Ένωση, ούτε από την Αφρική, γιατί ενδιαφέρουσαν οι συζητήσεις και για την ημερήσια διάταξη με την όλη η χορεογραφία και τα θέματα που θα συζητηθούν στα επόμενα προγράμματα δράσης. Σίγουρα ελπίζουμε και εμείς ότι και όλοι θα παίξουν ενεργό ρόλο στα πλαίσια της ε, Συνόδου Κορυφής. Και αυτό, όπως είδαμε, το ζήτησαν οι περισσότεροι που μίλησαν σήμερα. Τώρα, για τα επιμέρους θέματα. και εμείς κάπως ανησυχούμε για τη μειωμένη φιλοδοξία. Ξεκινήσαμε καλά στη Λισαβόνα, αλλά πρέπει να μεταφράσουμε αυτά σε συγκεκριμένη δράση. Και πρέπει να εστιαστούμε σε κάτι που να, δίνουν, να δίνει απτά αποτελέσματα. Σαφή προστιθέμενη αξία με περιφερειακή και παναφρικανική διάσταση. Αυτή είναι και η δική μας φιλοσοφία. Είμαι αισιόδοξο ως προς το ότι εν μέρη το πετύχαμε αυτό. Φυσικά θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα έχει να πει για τα επόμενα προγράμματα δράσης στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε τα Κοινοβούλια, όπως είπα, να παίξουν ενεργό ρόλο, όχι μόνο στην παρακολούθηση, αλλά και στην εφαρμογή, όπως η δημοκρατική διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν γίνεται χωρίς τα Κοινοβούλια. Ξανατονίζω ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για ανοιχτή συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν το θέλει αυτό. Το ίδιο ισχύει και για άλλους ε, μη κρατικούς φορείς. Θέλουμε και η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικό τομέα να παίξει πιο ενεργό ρόλο. σχετικά με το πώς θα ενισχυθεί το δυναμικό στην Αφρική, τα πρακτικά δηλαδή θέματα, συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας στην Παναφρικανική Ένωση, έτσι ώστε να αυξηθεί αυτό το δυναμικό, η πόροι. Φυσικά έχουμε δυσκολίες με το δίκτυο απορροφητικότητάς τους. Πάντως συνεργαζόμαστε. Αυτά προς στιγμή. Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο για να κλείσουμε. Ευχαριστώ για να δώσω και την ευκαιρία και στην γερμανική καμπίνα να κάνει ένα διάλειμμα. Λέει ο κύριο Γκάλερ, σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνώ απόλυτα ότι με αυτά που είπε ο κύριο Μπέρμαν ότι ο πλούτος ε, ο οποίος ε, δημιουργήθηκε στην Αφρική τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να κατανεμηθεί διαφορετικά και μάλιστα από αφρικανικής πλευράς εμείς δεν χρειάζεται να αναμειχθούμε αλλά αν μας το ζητήσουν σίγουρα θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες κατασυντήρες γραμμές για το πώς θα πρέπει να επιτευχθεί αυτό και στο ψήφισμα περιλαμβάνεται ένα σημείο ακόμα που αναφέρεται ότι η φοροδιαφυγή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια στις αφρικανικές κυβερνήσεις κάθε έτος. Δηλαδή τα έσοδα από το πετρέλαιο και από άλλες πρώτες δεν φαίνεται να ωφελούν όσο θα έπρεπε τα διάφορα κράτη. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα θέμα. Πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και θεωρώ ότι οι μη κρατικοί φορείς θα πρέπει να κατοχυρωθούν στις εταιρικές σχέσεις, στις σύμφωνες εταιρικής σχέσης. Ίσως θα έπρεπε να αναφέρονται ρητά. Δεν ξέρω πού ακριβώς ε, θα μπορούσαν πρακτικά να αναφερθούν, αλλά σίγουρα θα μπορέσαμε να βρούμε μία λύση. Η θεσμική ενίσχυση αποτελεί ένα θέμα που και εμάς μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ασφαλώς και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι δύσκολο γιατί δεν είναι απλό, ξέρετε, να το πετύχουμε αυτό για όσους άμεσα συμμετέχουν. Ωστόσο, είναι ευγενής ο σκοπός. Η συνοχή. Ίσως η συνοχή αυτή της πολιτικής, και το αναφέρω αυτό επειδή το είπατε, ίσως θα έπρεπε να αναφέρεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στο ψήφισμα. θα μπορούσαμε όντως να το έχουμε διατυπώσει κάπως καλύτερα. Κατά τα άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα χρόνια και για την ανοιχτή στάση που επέδειξε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλαμε και εμείς λοιπόν να ακουστεί η φωνή μας και από πλευράς μας επιθυμούμε να συνεχιστεί, να συνεχιστεί αυτό. Η κριτική που ανέφερα προηγουμένως δεν απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιθέτως, γιατί θεωρώ ότι η Επιτροπή και αυτή δυσαρεστείται όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση επαρκής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας θυμίζω οι προθεσμίε Τροπολογίες σήμερα το βράδυ σε 7 η ώρα. Πέρας. Ψηφίζουμε αύριο. Πρώτα θα το δουν οι συντονιστές. περνάμε στο σημείο 7. Φορολογία και ανάπτυξη. Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πρόθεση χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα. Είμαι η συγγήτρια της έκθεσης πρωτοβουλίας άρθρο 50 παρατηρητές, η ΕΚΟΝ και η ΙΝΤΑ θα γνωμοδοτήσει. Σήμερα είναι μια πρώτη παρουσίαση της έκθεσης. Θα συζητηθεί με τα έγγραφα στις 8 Νοεμβρίου, προθεσμίες 11 Νοεμβρίου και ελπίζουμε στις 18 Ιανουαρίου να ψηφίσουμε το κείμενο. Τώρα θα σα περιεργασιάσω σε γενικέ γραμμέ την έκθεση αυτή. Θα το πω στα αγγλικά. Επικροτούμε την πρόταση της Κομισιόν που μας δίνει ενισχυμένη βοήθεια για τη βοήθεια ανεπισόμενων χωρών σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση του φορολογικού συστήματος. Υπενίζομαι πόσο στενή είναι η φορολογητέα βάση σε αναπτυσσόμενες χώρες που υποφέρουν από εξαιρέσεις φορολογικής πίεσης προς τους πλούσιους και παράνομες ε, ροές κεφαλαίων σημειώνονται που έχουν σχέση με την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Οι υποχρώσεις του ΠΟΕ και οι περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες δημιούργησαν οξέα προβλήματα για τις πιο φτωχέ χώρες που αντικατέστησαν περίπου το 30% των χαμένων φόρων μέσω του εμπορίου που δεν μπορούν να τους αντικαταστήσουν με κάτι άλλο. Με την άμεση φορολογία προκειμένου. Επίσης, στο εγγραφό μου τονίζω το ότι υπάρχει ανισομέρεια μεταξύ της φορολόγησης των κατόχων κεφαλαίου και των μισθωτών. Αυτό θα έπρεπε, η ψαλίδα έπρεπε να μικρύνει. Μετά έχουμε την ε, κακή εμπορική τιμολόγηση. Η G20, ο ΣΑ, ε, η ΠΟΕ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πιο ευρύς δείκτες και μεθόδους για να αντιμετωπιστεί αυτή η κακή εμπορική τιμολόγηση. Θα πρέπει να δούμε τις ε, συγκριτικές μεθόδους που έχουν στις ΗΠΑ που υπόσχονται πολλά. Επίσης, καλούμε την Ένωση στους G20 και την ΟΣΑ να υποστηρίξει την αρχή της αυτόματης συνταλλαγής πληροφοριών στα φορολογικά, όπως έχουμε την οδηγία εμείς για τη φορολογία καταθέσεων είναι ο πιο καλός τρόπος να καταπολεμηθεί η παράνομη ροή κεφαλαίων. Η ποιότητα επίσης των εκθέσεων συλλογισμών κλπ. είναι απολύτως αναγκαία για τον φορολογικό έλεγχο και θα πρέπει να ισχύσουν οι διεθνή λογιστικά πρότυπα. Όλες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουν το, τα έσοδα και τον φόρο που πληρώνουν κατά χώρα. Δεν θα πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας για να ξεριζωθεί η παγκόσμια φτώχεια αν δεν πάρουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων και παράνομων φορολογικών υποδομών. Από τη διάσκεψη των G20 του Απριλίου του 2009, τα περισσότερα κέντρα offshore δεσμεύτηκαν να εφαρμογήσουν τις διεθνείς προδιαγραφές για τη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, ε, εξακολουθεί να ισχύει αυτή η δομή των φορολογικών παραδείσων και πρέπει να ξεπεράσουμε το πλαίσιο του ΩΣΑ για να κατεπολεμηθεί αυτή η ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων και η... τα προβλήματα που δημιουργούν. Έχω μία μικρή παράγραφο για τα ταχύς, ατυχείς επιπτώσεις στην διανομή των φορολογικών εισοδημάτων λόγω των συνθήκων. Ε, μάλλον διαφορών εμπορικών φορολογικών συμφωνιών και ο πιο καλός τρόπος να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή είναι να έχουμε μια διεθνή συνθήκη να πάψουν να υπάρχουν ε, φορολογικές δομές οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη υπάρχει η νομοθεσία του Stop Heaven Tax Abuse στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν ήσασταν στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματεία των ΗΠΑ Εθνών, τον Μπαν Κιμούν, όπου χρησιμοποίησε το χρόνο μιλίας που είχα δύο λεπτά και τον ερώτησα συγκεκριμένα. Αν θα προωθήσει μια διεθνή συμφωνία για φορολογικά θέματα. Δυστυχώς το έκανε αυτό στα γαλλικά και δεν ξέρω αν το... με κατάλαβε. Πάντω ζήτησε ένα ραντεβού να του εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και ελπίζω και πιστεύω ότι θα μου δοθεί αυτή η δυνατότητα για αυτή τη συνάντηση. Αυτά σε γενικές γραμμές η έκθεσή μου. Στις 8 Νοεμβρίου θα σας μοιραστεί. Μπορείτε να κάνετε και τροπολογίες μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Ο κύριος Ντάνσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ε, διαβάσω κάτι από τον Βολφ Κλίντς που είναι ο σχεδόν εισηγητή των φιλελευθέρων και γενικότερα εξ ονόματο των φιλελευθέρων. Επικεντρούμεθα όσον αφορά τι φορολογικέ ρυθμίσει τη αντισώμενη χώρα, τόσο ώστε να είναι δυνατόν να μην βλέπουμε στο τι έχει ε, ε, ξοδευτεί, αλλά τι έχει ε, εισπραχθεί, οπότε θα πρέπει ο στόχος να είναι αυτές οι χώρες να μπορούν να αυτενεργήσουν και ο οποιοδήποτε άλλος προβληματισμός σε εκείνες τις χώρες θα πρέπει να έχει αφετηρία το ότι ο προσωπικός φόρος εισοδήματο τελικά δεν αποδίδει σαν εισόδημα για αυτές τις χώρες, διότι πάρα πολλοί οι οποίοι υπόκειται σε αυτόν τον ε, είναι πάρα πολύ λίγη σε σχέση με τις βιομηχανικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, το να εισπράτεται ο φόρος φυσικά και προποθέτει να υπάρχει φορολογική βάση και κάποιες εταιρείε που να μπορούν να λειτουργήσουν στις χώρες αυτές και φερειπίν υπάρχουν πάρα πολλές ε, εταιρείε που ασχολούνται με εξόριξη πρώτων υλών, όμως πολλές φορές Έχουμε το παράδοξο τη ε, αυθονία στι χώρε αυτέ, γιατί είναι χώρε οι οποίε έχουν πάρα πολλού πόρου, όμω ε, έχουν αργό ρυθμό ε, ανάπτυξη σχέση με τι αναπτυσσόμενε χώρε τελευταία 40 ετία και ο ένα ε, χώρο για αυτό το μη οικονομικό λόγο είναι ότι αυτέ ε, οι χώρε δεν έχουν κανένα είδου φορολογικά έξοδα, μια που δεν υπάρχουν οι αρμόδιε φορολογικέ αρχέ ή γιατί οι εταιρείε στι χώρε αυτέ βγάζουν τα, τα, τα κέρδη σε άλλες χώρες με μικρότερους συντελεστές και γι' αυτό και η φορολογική, η φορολογική πολιτική δεν γίνεται όπως θα πρέπει. Ας πούμε η Βρετανία λέει ότι 35 δις ευρώ χάνονται και μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 100 δις αυτά τα οποία θα μπορούσαν ε, σε, στον, χώρε χώρες να εισπράττουν από τις ε, εκεί δρούσες εταιρείες οπότε θα πρέπει η ε, αναπτυξιακή πολιτική να μην είναι μόνο το να στηθούν τέτοιε φορολογικέ αρχέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και τιμιότητα για τα φορολογικά και να υπάρχει διαφάνεια κυρίω όσον αφορά τι πολυεθνικέ, τι χώρε εκείνε. Και αυτό με τη σειρά του προαπαιτεί ότι οποιαδήποτε φορολογική αρχή θα πρέπει να έχει εξουσίες κατάλληλες και να μπορεί να ελέγξει τις εταιρείε όπου και να δρούν αυτές, όπου και να έχουν έδρα και επίσης θα πρέπει να είναι δυνατόν να μην γίνονται κάποια λάθη όσον αφορά το φορολογικό σύστημα. Γιατί πολλές φορές τα φορολογικά συστήματα είναι περίπλοκα και δεν βοηθάνε σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες. Άρα ε, δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που γίνονται εδώ στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κεντρωθούμε στη, στη ισότητα και απλότητα όσον αφορά τα φορολογικά συστήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσμαν, έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόνσκης γιατί τα περισσότερα από όσα είπε θα τα έλεγα εγώ. Συμφωνώ 100%. Δεν θυμάμαι εξ ονόματος ποιου το διάβασε, πάντως συμφωνώ με το κείμενο. και αυτό μου θυμίζει το ότι παλαιότερα είχατε καλέσει κάποιον Αμερικανό, το οποίο το όνομα δεν θυμάμαι, ο οποίος είπε ακριβώς το ίδιο. Πριν από ένα χρόνο περίπου. Και επίσης τον ΟΗΕ, σε κάποια συνάντηση κορυφής των αναπτυσσομένων χωρών, είχε αναφερθεί αυτή η φυγή κεφαλαίων. εκ μέρους ευρωπαϊκών εταιριών που βγάζουν τα κέρδη για να πληρώσουν εκεί φόρα και τα στέλνουν σε φορολογικούς παραδείσους. Άρα πάρα πολύ σωστό αυτό το να επικεντρωνόμαστε στους φορολογικούς παραδείσους. Μέχρι την επόμενη διετία. Θα διαπιστώσουμε το πόσο κάποιες χώρες ευρωπαϊκές διστάζουν να κάνουν κάτι για τους παραφορικούς παραδείσους και γι' αυτό και εγώ νομίζω θα πρέπει να αποδείξουμε με έρευνα πόσα είναι τα χρήματα εκείνα τα οποία ξαναγυρίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις εταιρείες που, τα, που βγάζουν τα κέρδη έξω. Βεβαίω και πρέπει να γίνει καλύτερη διακυβέρνηση στα οικονομικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά έτσι κι αλλιώς όσον αφορά τι μειονότητες δεν έχουμε και πολύ σωστή διακυβέρνηση. Αυτό το ξέρετε, με λυπή κατάσταση. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή. Αλλά τι να την κάνουμε τη χρηστική διακυβέρνηση, αν δεν εισπάτονται φόροι. Χρειάζεται εκεί η σωστή διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να έχουμε προφάσεις. Θα πρέπει επομένως να εφαρμοστούν αυτά τα, αυτές οι προστάσεις για τη φορολογία και αυτό θα πρέπει να τα ξεκινήσουμε από τα του οίκου μας, από την Ευρώπη δηλαδή. Έχετε το λόγο κυρία. Ευχαριστώ για την έκθεση είναι, ε, βοηθάει, όπως είπε και το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Φορολογική Ακαιριότητα, που λέει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες κάνουν χώρα χάνουν 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τη φορολογία. Και αν σας κατάλαβα καλά, λέτε πρώτον να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά που είναι δυνατόν να διορθωθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει και αυτές να κάνουν κάτι προκειμένου η σχέση αυτή να γίνει πιο δίκαιη. Και ενώ υπάρχουν διαφεύγοντα φορολογικά έσοδα λόγω ημών με Χαίρομαι πολύ που μας δίνει τη ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση και σήμερα και αργότερα. Πρόεδρος, η Κομισιόν θέλει να μας πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θυμίζω το ρόλο που εσείς παίξατε σε σχέση με την ανακοίνηση της Κομισιόν για την φορολογία και την ανάπτυξη και την πρώτη συζήτηση που είχαμε δώσει στη διάρκεια της διαβούλευσης. Δηλαδή, έχουμε τις ίδιες ιδέες με σας, τους ίδιους στόχους. Η έκθεση αυτή έρχεται στη κατάλληλη στιγμή όπου για τη φορολογία την περισμένη εβδομάδα η Κομισιόν ενέκρινε την πράσινη βιβλίο για τα δημοσιονομικά, διότι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της διαβούλευσης για το δημοσιονομικό ΑΕΠ είναι η σχέση μας ανάμεσα στο δημοσιονομικό ΑΕΠ και η κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων. Αυτά για την πράσινη βίβλο. Για μας ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν ένα διαφανές φορολογικό σύστημα, ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα με δύο διαστάσεις. Την εσωτερική διάσταση, δηλαδή η φορολογική διοίκηση να μπορεί να εισπράττει τους φόρους και να έχει την κατάλληλη φορολογική πολιτική προκειμένου να αναπτυχθεί και ο ιδιωτικό τομέα αλλά και ο φορολογούμενος να μπορεί να συμβάλλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Και η δεύτερη διάσταση, η διεθνής. και όπως είπαν και οι ευρωβουλευτές που ήδη μίλησαν, η διεθνής διάσταση περνάει μέσα από έννοιες που εσείς, κυρία Πρόεδρε, αναφέρετε, έκθεση κατά χώρα, ανταλλαγή πληροφοριών και οι τιμές μεταφοράς, μεταβίβασης. με τους συναδέλφους μας, για το θέμα είναι περίπλοκο, εμείς από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης φροντίζουμε οι αποφάσεις της Κομισιόν να υπάρχει η διάσταση ανάπτυξη, αλλά έχουμε και θέματα εσωτερικής αγοράς, όπου οι συνάδελφοι της φορολογικής διεύθυνσης είναι πιο αρμόδιοι. Πριν από 15 μέρες ε, συστάθηκε μια ειδική ομάδα υπό την διεύθυνση της Διεύθυνσης Φορολογικών Θεμάτων και η ενθάρρυνσή σας είναι ευπρόσδεκτη και η Κομισιόν σε το χρόνο θα έρθει να συζητήσουμε την έκθεσή σας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο σημείο 9. χορήγηση της εγγύησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύηση για τα σχέδια εκτός της Ένωσης. Έχουμε ένα σχέδιο απόφασης για να ενισχυθεί η εξωτερική εντολή της ε, ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον πόρων. Βέβαια, η τροποποίηση αυτή τη εξωτερική εντολή επηρεάζει το ρόλο τη τράπεζα σχετικά με τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και επειδή η διάσταση ανάπτυξη του θέματο αυτού είναι σημαντική, ζητήσαμε βάσει το άρθρο 50 το καθεστώ τη συνδεδεμένη επιτροπή με την Επιτροπή Προεπολογισμού, που είναι η αρμόδια. Η διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε αυτό το αίτημά μας. Τις Μπέρμαν είναι ο συγητής μας για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης για την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι δεν μας δόθηκε το καθώς που ζητήσαμε βάσει τα άρθρα 50, έχουμε άριστη συνεργασία με τον εισηγητή Κάλφιν και είμαι σίγουρος ότι θα λάβει υπόψη σχεδόν όλες τις τροπολογίες μας. Και για να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα. Η εξωτερική εντολή της ΕΤΕΠ ε, έχει να κάνει κυρίως με αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή όχι μόνο σε χώρες γειτονικέ, αλλά και σε πιο μακρινές αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό έχει συνέπειες, θα πρέπει μάλλον να αντικατοπτρίζεται και στο κείμενο της εξωτερικής εντολής. Θεωρώ ότι η καταπολέμηση της ένδυας θα πρέπει να αναφερθεί ρητά στην εντολή της τράπεζας. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι δεν χρειάζεται να αναφερθεί ρητά, γιατί και η ΕΤΕΠ θα πρέπει να τηρεί την στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τονιστεί πιο ρητά. Άρα αυτό θα αποτελέσει σίγουρα μία τροπολογία, την οποία ευχαρίστως θα δεχτούμε. Θα πω και κάποια άλλα σημαντικά θέματα. Θα πρέπει η ΕΤΕΠ να ενισχύσει ε, project στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, τα οποία επηρεάζουν πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά και την πιο εύκολη ε, ε, πρόσβαση για σε πιστώσεις από άτομα τα οποία παραδοσιακά έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση, όπως οι γυναίκες, όπως οι εθνικές μειονότητες. γιατί πολλές φορές οι τράπεζες θεωρούν ότι δεν είναι αξιόπιστα, δεν έχουν φερεγγιότητα αυτές οι ομάδες. Αλλά το 80% για παράδειγμα των αγροτών είναι γυναίκες. Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τα ταμιευτικούς λογαριασμούς, πιστώσεις και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ αργή η ανάπτυξη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν ο ρόλος της ε, ΕΤΕΠ να είναι η ενίσχυση, η αλλαγή της κατάστασης αυτής, η ενίσχυση αν θέλετε των μικροπιστώσεων και των αγροτικών τραπεζών. Μία επιπρόσθετη πτυχή της εντολής της ΕΤΕΠ είναι η διοχέτευση πόρων σε μέσα περιβαλλοντικά. αρκεί να διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για κονδύλια τα οποία προέρχονται από το κανονικό προπολογισμό της ΕΤΕΠ για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θεωρώ ότι η ΕΤΕΠ μπορεί να συμβάλλει περισσότερο και πιο έντονα ως κινητήριος μοχλός για τη συνεργασία, για τη συνεργασία μάλλον την διμερή συνεργασία με άλλες τράπεζες όπως ε, ολλανδικές ή γαλλικές τράπεζες Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και στο σημείο αυτό θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί πιο έντονα η ΕΤΕΠ, να υπάρχει πιο έντονη προσπάθεια να καταβάλλεται από τις διάφορες εθνικές ε, τράπεζες. Όλα αυτά φυσικά προϋποθέτουν ότι θα υπάρχει πιο πολύ προσωπικό και αυτό είναι μια ανάγκη την οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Δεν χρειάζεται πολλά άτομα, αλλά θα πρέπει να έχει τους επαρκείς πόρους η ΕΤΕΠ. Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση, ωστόσο, στην αναθεώρηση της εξωτερικής εντολής της τράπεζας είναι σωστή στη στιγμή να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες της τράπεζας σε ό,τι αφορά τα θέματα διαφάνειας. Η ΕΤΕΠ θα πρέπει φυσικά να τηρεί απόλυτα τον ε, δοντολογικό κώδικα που την διέπει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα έσοδα των project που υποστηρίζει, σε ό,τι αφορά τους φόρους, για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά το άχθος και πώς ε, κατανείμεται στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η κοινωνική και η αναπτυξιακή πτυχή. Και Επίσης, στις εκθέσεις που υποβάλλει, θα πρέπει να αναφέρεται κατά πόσον υπάρχει συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στις ε, εκάστοτε χώρες. Επίσης, στην ετήσια έκθεσή της, να το πω θα πρέπει να υποβάλει ετήσιες εκθήσεις η ΕΤΕΠ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις πτυχές της ε, εξωτερικής εντολής. Γιατί αυτό θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που τύφονται ως προς τη διαφάνεια και ως προς τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μίτσελ. Α, δεν ζήτησε το λόγο ο κύριος Μίτσελ. Εντάξει, λοιπόν. Monsieur Newton. Voilà. Monsieur Newton. Όπως είπε και ο κύριος Στέις, ε, δεν μπορώ να έρθω στις 6.30 στη συνάντηση, αλλά θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε απόλυτα τις προτάσεις του. Σας βοηθάει αυτό? Ναι. Ωραία, ναι, ναι, ναι με βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά ακύρωσα την συνάντηση αυτή γιατί κανείς δεν μπορούσε να έλθει. Θα πάρω τώρα τον, τον λόγο και ευχαριστώ τον κύριο Μπέρμαν για το έργο που επιτέλεσε όσον αφορά την αλλαγή της εντολής. Θα πρέπει να τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αποτελούν η φορολογική παράδειση, γιατί θα πρέπει να πετυχθεί από τις εταιρείε ε, οι οποίες την χάνουν τέτοιων χορηγήσεων να τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τον ε, φόρο στο, στο στα κέρδη και ε, παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι δεν έχουμε θίξει το ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παραπομπή στη συμφωνία του 2005 της Κοπενχάγης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αναπτυσιακής βοήθειας. Θα πρέπει δε η χρηματοδότηση να έχει προτεραιότητα ούτως ώστε να επιλεχθούν οι στόχοι της χιλιετίας. Επίσης, πρέπει ε, οποιοδήποτε πρόγραμμα να είναι συμβατό με την αλλαγή του κλίματος, να έχει καθαρή τροπολογία, οπότε με την αδειά σας θα υποβάλλω τις σχετικές τροπολογίες. Μήπως θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κασόνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μπέρμαν. Νομίζω ότι η δουλειά του και η προπαρασκευαστική δουλειά που έγινε με τη μελέτη είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και έτσι βελτιώνει την ε, δουλειά μας σε σχέση με αυτή την ε, εντολή και νομίζω ότι η ίδια η Επιτροπή έχει προτείνει να γίνει προοδευτικά ε, μεγαλύτερη η συμβολή της ΕΤΕΠ Αυτό όμως προοδευτικά, ή δεδάλλως, Η δάλος, η πραγματικότητα θα μας προσγειώσει απότομα. Γιατί όντως μπορεί να βοηθήσει για την οξιακή βοήθεια η ΕΤΕ και τη τα πολέμηση της ε, φτώχειας. Όμως σήμερα είναι δύσκολο αυτό να το έχει ως κύριο στόχο η τράπεζα. Όπως είπε ο κ. Μπέρμαν, πάμε για το 2014 και πέρα για αυτή τη δουλειά. Άρα, όσον αφορά αυτή την εντολή, θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πιο προσεκτική. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει υποχρέωση ε, λογοδοσίας, υποπτία, παρακολούθηση κατά όλη τη διαδρομή, όπως τα είπε και ο κύριος Μπέρμαν. Τώρα, όσον αφορά τα offshore τα κέντρα δραστηριότητα. βεβαίως και θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια αλλά θα πρέπει να είναι δυνατόν η τράπεζα να ασκεί μια πολιτική που να συμμορφώνεται με τα όσα θέλουμε και εμείς αλλά θα πρέπει να συμμορφώνεται και με του κανόνε λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τα σχετικά προγράμματα. Και συμφωνώ με όλε τι αλλαγέ που προτείνει ο κύριος Μπέρμαν. Και τώρα για την ΕΤΕΠ, ο κύριος Καρανό έχει το λόγο. Merci beaucoup. Euh, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπέρμαν για την έκθεση και για την τόσο καλή συνεργασία. Για το πόσο προσπαθεί να βελτιώσει την εντολή. Έχω μια-δυο παρατηρήσεις. Πρώτα από εδώ όσον αφορά την ε, αναπτυξιακή συνεργασία πρόκειται για την καρδιά της εντολής. Και αυτό τώρα αντιστοιχεί στην νομική βάση που έχουμε για αυτή τη συνεργασία που είναι πολύ σημαντικό. όμως θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Τι ζητείτε από την ΕΤΕΠ να πράξει και από την άλλη μεριά από τον τρόπο λειτουργίας στη δομή της ε, ΕΤΕΠ. Όπως ξέρετε η ΕΤΕΠ ε, έχει πολύ λιγότερο προσωπικό από ότι άλλα τέτοια, άλλες τέτοιες υπηρεσίες, άλλες τέτοιοι φορείς, άλλες τέτοιες τράπεζες. Άλλε τράπεζε δηλαδή που έχουν εγγραφεί τη δουλειά τη ανθρωπιστική βοήθεια και τη κατανόηση τη φτώχεια ω κύριο στόχο. Άρα, εάν θέλουμε η ΕΤΕΠ να βοηθήσει περισσότερο για του στόχου μα, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπο λειτουργία τη ΕΤΕΠ όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων εκτός ΕΕ. Βαθμία η Κομισιό θα πρέπει να είναι η προσέγγιση, να ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση των μελετών των επιπτώσεων και όσον αφορά αυτά τα χρηματοοικονομικά κέντρα, τα offshore, Βεβαίως θα πρέπει να προσέξουμε τις ε, απάτες, τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και γι' αυτό κάθε κίνηση τέτοια είναι ευπρόσδεκτη. Το Συμβούλιο έχει πει ότι αυτό είναι βασικό κριτήριο για τα σχετικά προγράμματα. Πολλέ φορέ βέβαια θα πρέπει να σε συγχρηματοδότηση με κάποιου οργανισμού οι οποίοι δεν έχουν την ίδια αυστηρότητα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δυνατόν εμεί να ανεχθούμε την ε, αθέμητη χρήση των πόρων που χορηγούμε. Το για τους επίσημους καταλόγους δεν έχουμε εμείς εντολή και αρμοδιότητα να καταρτίζουμε καταλόγους χωρών ε, γι' αυτό και προσφεύγουμε στους καταλόγους που κάνουν άλλοι οργανισμοί, αλλά ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να το κάνει. Monsieur Berman, vous avez la parole pour conclure. Κύριε Σπέρμαν, για να ολοκληρώσει. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις και τις τροπολογίες που προτείνετε. Αν ε, καταλαβαίνει σωστά το θέμα. Δεν είναι δύσκολο να τι συμπεριλάβουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ απλέ και θα μα δουν σύμφωνου κάποιε από τι παρατηρήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. καταρχά, να σα ευχαριστήσω για τα σχόλιά σα για την προσέγγιση που προτείνετε. Ναι, όντω. Ασφαλώς, αλλά δεν νομίζω ότι η εξωτερική εντολή θα πρέπει να συμβαδίζει σε ό,τι αφορά την διατύπωση με την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει, αν θέλετε, μη ρητά. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ε, προδιαγραφές από την ε, συνθήκη, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι για λόγους αφήνειας, δηλαδή να διευκριστούν ρητά και στην εντολή της ε, ΕΤΕΠ. Πολύ χρήσιμο το σχόλιο σας από τον εκπρόσωπο της ΑΤΕΠ ότι λειτουργεί η τράπεζα με 10 φορές πιο λίγο προσωπικό σε σχέση με άλλα όργανα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ε, για τα άλλα όργανα δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με λιγότερο προσωπικό, αλλά σίγουρα εσείς χρειάζεστε πιο πολύ προσωπικό σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των χωρών τώρα, των αναπτυσσόμενων χωρών. Νομίζω ότι είναι ο κατάλογος του ΩΣΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci. Donc, je vous rappelle... Ευχαριστώ πολύ. Σας θυμίζω προθεσμία για τις τροπολογίες 26 Οκτωβρίου, 18 η ώρα και η ψήφο στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 9 ε, Νοεμβρίου. Και περνάμε στο 10. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων δεσμολογικών προτιμήσεων. Είμαι συγκήτρια για την γνωμοδότηση. Το σύστημα ΓΔΠ της Ένωσης είναι ένας εμπορικός μηχανισμός που επιτρέπει στην Ένωση να προσφέρει σε αναπτυσσόμενες χώρες προτιμησιακή πρόσβαση και μία αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές με μείωση των δεσμών. Το τρέχον σύστημα γάμα ορίζεται από ένα κανονισμό του Συμβουλίου που θα λήξει τέλος 2011. Από τώρα έχουμε ένα νέο σύστημα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί νομικό κενό. Η Κομισιόν θα υποβάλει νέα πρόταση αρχές του 2011 που σημαίνει ότι το νέο σύστημα ΓΔΠ θα ισχύσει περί τα μέσα του 2012 έξι μήνες μετά την λήξη του τρέχοντος συστήματος. Η πρόταση εδώ έχει στόχο να παρατείνει το τρέχον σύστημα ΓΔΠ για δύο χρόνια μάξιμουμ, μέχρι ότου ισχύσει ο νέος κανονισμός. Είναι καθαρά τεχνική πρόταση. Ωστόσο, ως εισηγήτρια για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, που θα τη στείλουμε στην ΙΝΤΑ, σκοπεύω να προτείνω και ορισμένε τροπολογίες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη και την πληροφόρηση του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να παρακολουθεί από πολύ κοντά την ουσιαστική αναθεώρηση που προβλέπεται για το 2011. Έχετε το λόγο. κανείς η Κομισιόν. Η κυρία Ιβόνα Ιτσικόφσκα, Κομισιόν. Όπως βλέπετε, δεν είμαι η κυρία Ιβόνα Ιτσικόφσκα λέω ο μιλητής που συνάδελας. Λέγομαι Μπέρες. Είμαι ο προϊστάμενης της κυρίας Τσικόφσκα. Πολύ σωστά τα είπατε. Πρόκειται για μία τεχνική πρόταση για να μην υπάρξει κενό. Και η θεμετή στόχη του συστήματος ΓΔΠ να τηρούνται και να μην υπάρξει αυτή η τεχνική δυσκολία. Αυτό που θέλουμε από εσά είναι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας επειδή πολλά σημαντικά θέματα διακυβεύονται και έχει σχέση λίγο και με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Πρέπει να δημοσιεύσουμε τον κανονισμό έξι μήνες πριν αρχίσουν να ισχύουν έτσι ώστε οι διάφοροι φορείς να μπορούν να προγραμματίζουν τη δράση τους. Που σημαίνει καλοκαίρι του 2011. Και ενδεχόμενοι νέοι υποψήφοι του συστήματος να υποβάλουν τις αιτήσει τους γνωρίζοντας με ποιο νομικό πλαίσιο θα δουλεύουν. Γιατί τα αιτήματά τους πρέπει να υποβληθούν πριν τις 31 Οκτωβρίου του 2011. Άρα και αυτοί μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να ξέρουν ποιοι όροι θα ισχύουν. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του κανονισμού ΓΔΠ το πλήρες εύρος της συμμετοχής του Κοινοβουλίου θα τύχει απόλυτου σεβασμού. Και όταν θα έχουμε το νέο κανονισμό, θα ισχύουν φυσικά οι όροι της συνθήκης της Λισαβόνας. Πλήρως. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. σημειώνω ότι συμφωνούμε να παρατεθεί το σύστημα ΓΔΠ που ισχύει σήμερα για να πάρουμε μέρος ενεργά στη συζήτηση για τον νέο κανονισμό. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία για τροπολογίες 26 Νοεμβρίου, 18 η ώρα, θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στις 9 Νοεμβρίου. Η ίντα θα ψηφίσει την έκθεση την 1η Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, θα διορθώσω κάτι, ένα λάθος έκανα. Ήθελα να πω 26 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία 19 Νοεμβρίου. Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα λύγουν, οι προθεσμοί για τροπολογίες. Έχουμε κερδίσει μία ώρα από τις εργασίες μας. Θα ψηφίσουμε. Και είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε στις 6 και 4. Προσωρινή διακοπή της συνεδρίασής μας μέχρι τις 6 και 4. όπου θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Κάσμαρεκ.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 nous Θα euh, euh, ψηφίσουμε στην γνωμοδότηση για κοινωνικές προδιαγραφές, κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα της Διεθνής Εμπορικές Συμφωνίες. Κύριο Κάσμαν, τροπολογία της Ζήμερ. κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Αποχές. Κατά, συγγνώμη. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Σαρτζεντίνιο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τέσσερα Σχέση με υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε, Σαρτζεντίνη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπάρχει αντίρρηση. Τότε ψηφίσουμε τη συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι της κυρίας Ζήμερ υπέρ, χωριστή ψηφοφορία. Ωραία, το πρώτο είναι τότε. Υπέρ, κατά, αποχές ξαναρχίζουμε υπέρ έξι Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Δέκα, ζήμερα, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Έντεκα, Σαζεντίνη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. οι 14-15 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψήφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην συγκεκριά. Αύριο συντονιστές σε νέα.